και το Ισραήλ θα συνοδευτούν από, την, από τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όχι από τη δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σημείο 3. αμέσως μετά τη συζήτηση της έκθεσης Goldstone για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη θα προσθεθεί ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη, η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής ε, για θέματα κοινωνίας των πολιτών και εθνικών μειονοτήτων στην Λευκορωσία. Η ψηφοφορία για το θέμα αυτό θα γίνει το Μάρτιο. Τέταρτη αλλαγή. Αμέσω μετά τι παρεμβάσει ενό λεπτού θα προσθεθεί το εξή σημείο στην ημερήσια διάταξη. Δήλωση τη Επιτροπή για μια σημαντική θεομηνία για την τραγική καταιγίδα που έγινε στην αυτόνομη περιοχή της Μαδέρας. Η ψηφοφορία για το σημείο αυτό θα γίνει επίσης το Μάρτιο. Ημέρα Πέμπτη. Τρία σημεία, τρεις αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Σε ό,τι αφορά την έκθεση Πατράων Νέβες για την κοινή ελευτική πολιτική, θα δοθούν πέντε λεπτά στο Συμβούλιο χρόνος αγόρευσης. Δεύτερη αλλαγή μετά τη συζήτηση της έκθεσης Πατράων θα προσθεθεί το εξής σημείο. Η δήλωση της Επιτροπής για θέματα ασφάλειας στις σιδηροδρομικές μεταφορές ε, συμπεριλαμβάνουν του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, Σηματοδότησης, χωρίς ψήφισμα και τρίτη προτινόμενη αλλαγή. Οι ψηφοφορίες θα αρχίσουν στις 11.30 αύριο, ημέρα 5η, 25 Φεβρουαρίου. Οι ψηφοφορίες θα αρχίσουν στις 11.30. Σε ό,τι αφορά την ε, Πέμπτη, η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέβαλε έτοιμα η ψηφοφορία της έκθεσης Λένε για τους ετήσιους λογαριασμούς σε ορισμένες ε, εταιρείε για μικροενότητες να αναβληθεί. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Σούλτς για το αίτημα αυτό των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, στην ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών ε, συζητήσαμε πάρα πολύ έντονα την έκθεση Λένε σήμερα το πρωί. Ναι, πάντα υπάρχουν ε, ενστάσεις. Gut. Ich fange nochmal von vorne. Να ξαναξεκινήσω λοιπόν, Πρόεδρε. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την διερμηνία. Με καταλαβαίνετε τώρα. Με ακούτε. Αφού με καταλαβαίνει και ο συνάδελφο Τσίστερ, Εντάξει. άλλο, λοιπόν, Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί λοιπόν η ομάδα μα έκανε μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση για την έκθεση Λένα και στην ομάδα μα. Δεν ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Αυτό συμβαίνει, ξέρετε, στις ομάδες, αλλά υπάρχουν υπάρχει επιθυμία να εκφράσουμε προς τον κύριο Λένε, τον εισηγητή, την επιθυμία να ξανασκεφτεί μέχρι τον Μάρτιο ποια πορεία θα χαράξουμε ε, σε ό,τι αφορά την εκθέση αυτή ως σοσιαλδημοκράτες. Από ό,τι ξέρετε υπάρχουν διάφορες ε, ε, απόψεις στην ομάδα μας. Αν λοιπόν θα γίνει αυτή η συζήτηση για να διαμορφωθεί η τοποθέτηση της ομάδας μας, νομίζω ότι καλύτερα θα βλεθεί μέχρι το Μάρτιο η ψηφοφορία. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε και εμάς αλλά και τις άλλες ομάδες για τη σχηματισμό άποψης. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε το λόγο για να υποστηρίξει αυτό το αίτημα. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο υπέρ του αιτήματος των σοσιαλιστών. Ο κύριος Λένε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι είναι καλό το γεγονό ότι οι σοσιαλδημοκράτε τόσο έντονα ασχολούνται με το θέμα αυτό. Αλλά διαπιστώνω ότι ω Κοινοβούλιο το Δεκέμβρη του 2008 σχεδόν ομόφωνα εξεδώσαμε ένα ψήφισμα στο οποίο καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση ακριβώ όπω αυτή που την οποία κοιτάμε τώρα. Λοιπόν, το Κοινοβούλιο κάποια στιγμή θα πρέπει να τηρήσει αυτά που αποφάσισε αυτά που αποτελούν πολιτική βούληση του οίκου μα εδώ και χρόνια. Φυσικά, σε κάθε νομοθετική πρόταση υπάρχουν κάπου αμφιβολίες και ερωτηματικά. Αυτά τα ανοιχτά ζητήματα τα επιλύσαμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων με συμβιβασμού. Αυτοί οι συμβιβασμοί είναι όριμοι για να περάσουν σε ψηφοφορία. Φυσικά μπορεί να υπάρχει κάποιο σκοπό, κάποια έννοια να συζητηθούν περαιτέρω, αλλά αν σκοπός του κυρίου Σούλτς είναι να απολαύσει μεγαλύτερη υποστήριξη σε η πρόταση αυτή. Δεν έχω αντίρρηση να αναβληθεί η ψηφοφορία μέχρι τον Μάρτιο. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε στους σοσιαλιστές την δυνατότητα, τη δυνατότητα να σκεφτούν την θέση που θέλουν να κρατήσουν σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις αυτές. Ποιος θα ήθελε το λόγο κατά του αιτήματος. Ο κύριος Στέρεξ, ευχαριστώ τον κύριο Λένε για τις δηλώσεις του, αλλά θα ήθελα να ζητήσω το εξής. Υπό τους όρους αυτούς, υπό τις συνθήκες αυτές, θα πρέπει να ζητήσω να γίνουν και τροπολογίες και συζήτηση, γιατί τώρα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, δεν υπήρχε δυνατότητα υποβολής τροπολογιών, προβλεπόταν μόνο η ψηφοφορία. Ο Πρόεδρε, να επαναλάβω αυτό που είπα. Φυσικά είμαστε υπέρ της συζήτησης, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να αναβληθεί η ψηφοφορία και θα πρέπει να πω για λόγους ε, δικαιοσύνης ότι καταλαβαίνω την επιθυμία του συναδέλφου λένε, αλλά στην ομάδα μας ε, κύριε Λένε επικρατεί δημοκρατία. Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Ας ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης της ομάδας σοσιαλιστών. Παρακαλώ, διανατάσσεω της χειρός ποιος είναι υπέρ της πρόταση των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Κατά. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται η πρόταση. Οπότε η ψηφοφορία της έκθεσης λένε για τους ετήσιους λογαριασμούς ορισμένων εταιριών σε ό,τι αφορά κάποιες μικροενότητες αναβάλλεται. Δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, οπότε οριστικοποιούμε το σχέδιο μερίσης διάταξης και το εγκρίνουμε. Ο κύριος Βόμποτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Τις τελευταίες δύο ημέρες, τις τελευταίες ημέρες μάλλον, έγιναν σημαντικές κινήσεις εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ηνωμένων Πολιτειών και του ειδικού απεσταλμένου του στο Αφγανιστάν. Και οι δύο αυτές ενεργείες είναι αμφιλεγόμενες και γίνονται διάφορες συζητήσεις. Δεν θέλω να επισέλθω σε στρατιωτικά θέματα, αλλά Πρόεδρε θα ήθελα να παρακαλέσω να έρθουν και στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να γίνει ε, σχετική συζήτηση και ελπίζω να μας υποστηρίξουν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Το λαμβάνω υπόψη. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020. Ενέργεια στη συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου του 2010. Πρώτος θα λάβει το λόγο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Χέρμαν Van Rompuy. Θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για την παρθενική ομιλία του Πρόεδρου Βαν Ρομπόη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια. Είναι η πρώτη σας ομιλία, κύριε Πρόεδρε, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε συμφωνήσαμε να σας δώσουμε περισσότερο χρόνο, γιατί ο κύριος Πρόεδρος θέλει να σας εκθέσει τις απόψεις του και για άλλα θέματα και θεσμικά κατά την